να ξεκινήσουμε με την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Να καλέσω την κυρία Φωτίγκα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, η ανθρωπιστική κατάσταση και η κατάσταση ασφάλειας στην κεντροαφρικανική δημοκρατία εξακολουθούν να είναι τραγικές και μάλιστα υπάρχει και επιδείνωση. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η μεταβατική, ε, στέφθηκε με επιτυχία και αυτό το αναγνωρίζουν ε, και οι κεντροαφρικανοί. Βέβαια φαίνεται ότι κράτησε πολύ λίγο αυτή η αποστολή εξαιτίας προβλημάτων της λειτουργίας της αποστολής μηνούσκα το ΙΕ. Τελικά η δική μας αποστολή δεν κατάφερε να διεκπαιρεώσει αποτελεσματικά την εντολή της. Και Παρ' όλα αυτά, χάρη στον ε, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τις προσπάθειες που γίνονται, ε, θα ενδύνει τις προσπάθειες της διεθνής κοινότητα και θα στηρίξει και την Αφρικανική Δημοκρατία, γιατί πραγματικά γίνεται αιστεία δραματικής ριζοσπαστικοποίησης και η επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας ε, είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεύτερο συντάκτη του ψηφίσματος, ο κύριος Λουί Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η εκεχηρία του Απριλίου του 2015 και το Εθνικό Συμβούλιο του Μπαγκή τον προηγούμενο Μάιο για την επανασυμφιλίωση, για τον αφοπλισμό ε, και τον επαναπατρισμό επιτρέπουν τη δημιουργία μιας πραγματικής ε, πολιτικής προοπτικής. Ε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και πάλι τη Γαλλία για την δέσμευσή της. Περιμέναμε μεγαλύτερη ελληνική από τις υπόλοιπες κοινοτικές χώρες ε, για την Κεντριοαφρικανική Δημοκρατία. Θα ήθελα επίση να συγχαρώ την κυρία Σάμπα Πάνσα και τι μεταβατικέ αρχέ για την αποφασιστικότητά του να διεκπαιρεώσουν τη διαδικασία αυτή. Και στι 3 Ιουνίου θεσπίστηκε ο νόμο για τη σύσταση του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου. Το Εθνικό Συμβούλιο μάλιστα υιοθέτησε το μεταβατικό σχέδιο συντάγματο που θα υποβληθεί εντό λίγου σε δημοψήφισμα. Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής μου είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ελεύθερες, αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές πριν τα τέλη του έτους. Δηλαδή να τηρήσουμε πιστά και αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Κοράου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι η ε, αντιπαράθεση που μπορεί να κλιμακωθεί σε εμφύλιο πόλεμο και είναι μια από τις πολλαπλές περιπτώσεις της Αφρικής, κράτους της Αφρικής που ένα κράτος πλουσιότατο σε φυσικούς πόρους που θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να έχει οικονομική μένει δεσμευμένο υποδουλωμένο σε μια διαφορετικού είδους απεικιοκρατία. διότι η επίσημη απεικιοκρατία της Γαλλίας έχει πάψει όμως έχει ξεκινήσει η οικονομική υποδηγέτηση ιδίως ό,τι αφορά την αγορά ξυλίας θα μπορούσαμε εδώ να ε, ε, καταγγείλουμε οφείλουμε τις ε, ασυνέπειες των δικών μας πολιτικών. Διότι από τη μια παρουσιάζουμε τις ιδέες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμη σήμερα καταγράφουμε κανόνες για την εξαγωγή ξυλίας και ε, βεβαίως ε, αυτό είναι στην πηγή πολλών συγκρούσεων. Ευχαριστούμε κύριο Παντζέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόσφατη κλιμακοσυμβία μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων τη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι κάτι που μας ανησυχεί. Και αυτή η επιδείνωση της κατάστασης είναι ένα από τα πολλά επεισόδια της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή από το 2012. Τα τελευταία τρία χρόνια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχουν διαπραχθεί εγκλήματα σοβαρότατα συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν για το σκοπό αυτό, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, να παρέμβουμε με τρόπο σαφή. Χρειάζεται ένα εύρυθμο δικαστικό σύστημα λόγω χάρη που να ε, διεξαγάγει ε, ενδελεχείς έρευνε για όλε τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. Θα πρέπει ε, οι αρχέ τη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποθήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσει για να βοηθήσουν ακριβώ αυτή την κυβέρνηση να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση κρίση και να μεταβεί προ ένα νέο καθεστώ που να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων και να είναι δημοκρατικό. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρο. ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι νέε συγκρούσει του Σεπτεμβρίου αποδεικνύουν πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ανησυχώ από την ε, αναβίωση των ε, συγκρούσεων. Το Σάββατο μας πέρασε πυρπολήθηκαν δύο χριστιανικές εκκλησίες υπήρξε απόπειρα δολοφονίας ενός χριστιανού ηγέτη. Οπότε το βασικότερο είναι να περιοριστεί η βία και να επιστρέψει η χώρα στην διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, κράτους δικαίου και των εκλογών. Δεν είναι δυνατόν ε, χριστιανοί να μάχονται τους μουσουλμάνους. Ε, π.χ. συχνά ε, μία ένοπλη ομάδα θεωρείται χριστιανική παρά το ότι ε, στην πραγματικότητα δεν πιστεύει σε τίποτα. Ε, χρειάζεται λοιπόν, όπως είπαμε, πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια και να διεξαχθούν κανονικά εκλογές. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σύγκρουση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία μαζί με αυτήν στο Σουδάν και τη Συρία είναι μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Αλλά βέβαια αυτή στην κεντροαφρικανική δημοκρατία την έχουμε ξεχάσει. Οι αντάρτες ε, στην χώρα αυτή κάνουν ε, απαγωγές, ε, εκτελέσεις, και βεβαίως ε, η χώρα χρειάζεται βοήθεια αλλά ο Ερυθρός Σταυρός δεν μπορεί καν να πάει στην ε, χώρα ούτε στην πρωτεύουσα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οι ασθενείς πάνε με τα πόδια άμα βρουν ε, ιατρία οι αντάρτες πολεμούν και τους κιανόκαρνους και πληρώνουν τους άντρες τους με διαμάντια και σκληρή ξυλία. Και βεβαίως ε, ο καθένας κρύβει τα προϊόντα, τα διαμάντια δηλαδή και δημιουργούνται έτσι από θέματα τα οποία θα ξαναεμφανιστούν μόλις υπάρξει ειρήνευση. Και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αγοράζουν αυτά τα διαμάντια και την σκληρή ξυλία και βέλγικες επιχειρήσεις επίσης. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν αμέσως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να στερήσουν την χρηματοδότηση από τους αντάρτες. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Βεριζιά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αντιμετωπίσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της. Όλος ο πληθυσμός έχει πληγεί, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μισός σχεδός πληθυσμός και πολλά παιδιά μεταξύ αυτών ε, χρήζουν άμεσης ε, ε, βοήθειας ανθρωπιστικής και επισητιστικής. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την προοπτική μας εδώ. Έχουμε πολιτικοστρατητικές ομάδες που προσπαθούν να καπηλευθούν τους πόρους, ε, διαμάντια και ξυλία, με την συνενοχή των μεγάλων πολυεθνικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα απ' όλα σε μια πολιτική και όχι στρατιωτική επίλυση της σύγκρουσης και να χτυπήσουμε τις, ε, το, τις ρίζες του κακού, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά πρώτα απ' Επίσης, ε, ισχυρισμοί ε, για την διάπραξη εγκλημάτων από την ε, γαλλική στρατική επιχείρηση του Σαγκάρης θα πρέπει να διερευνηθούν. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Χαιρόμαστε για τις προσπάθειες που θα γίνουν εκλογές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει οι προσπάθειές μας και πολύ αμφιβάλλουμε αν θα διεξαχθούν εκλογές υπό κατάλληλες συνθήκες. Ευχαριστώ κύριος Βέντα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Και μάλιστα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική της κρίση από την ανάκτηση της ανεξαρτησία της. Και μάλιστα οι εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών έχουν φτάσει σε έξαρση, υπάρχουν εσωτερικοί εκτοπιστέντες, η κατάσταση ανθρωπιστική είναι κατεπίγουσα. Βέβαια ενισχύσαμε την ε, οικονομική μας ε, υποστήριξη ε, και χρηματοδοτούμε όχι μόνο ανθρωπιστικά σχέδια αλλά και αναπτυξιακά ένταξη των γυναικών στο, στο, στην αγορά εργασίας, προγράμματα υγείας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, όμως ε, πρώτα απ' όλα να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξηθεί η ασφάλεια στη χώρα αυτή. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες. Ο κύριος Ζιλ Παρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, φαίνεται... Ε, 61 νεκρούς είχαμε, 300 τραυματίες την περασμένη εβδομάδα στο Πανκί. Πάλι κλειδονίζεται η ειρήνη στη χώρα αυτή. Είχαμε υποβάλει προτάσεις για τον Μπανκί που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες κύριε Πρόεδρε θα πρέπει πρώτα απ' όλα και εντάχει να οργανώσουμε τις νομοθετικές εκλογές γιατί η, μεταβατική αυτή, η πολιτική αυτή μετάβαση δεν υπάρχει πια όπως είχε επιθυμήσει η πρόεδρος, η μεταβατική πρόεδρος Σάμπα Πάνσα. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις νομοθετικές εκλογές και ε, κυρίως ε, να επιταχύνουμε τη διαδικασία αφοπλισμού των πολιτοφυλακών και να προετοιμάσουμε το μέλλον ε, ενισχύοντας τη σταθερότητα. Μάλιστα, ε, έχουμε το φόρουμ του Μπανκί με 74 εκατομμύρια για το μέλλον της χώρας, αλλά δεν αρκούν 74 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε δραστήριοι, ενεργητικοί και όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και να τροφοδοτήσουν αυτό το ταμείο. Η κυρία Σένερα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι η λαιλασία των φυσικών πόρων είναι η αιτία της εξαθλίωσης και της φτώχειας σε ολόκληρη την Αφρική. Στην περίπτωση της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας γνωρίζουμε το συμφέρον των πολυεθνικών εταιριών για το πετρέλαιο, την ξυλία και τα διαμάντια. Με βάση τα στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι μεγαλύτερε εταιρείε ξυλία και πολύτιμων λίθων συμμετείχαν ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον εξοπλισμό των ένοπλων δυνάμεων, σε συνοπτικέ εκτελέσει, σε βιασμού, σε εξαφανίσει. Διερωτώμε λοιπόν, μέχρι πότε θα επιτρέπουμε αυτή τη λαιλασία των φυσικών πόρων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μέχρι πότε ή μάλλον πότε θα θέσουμε τέρμα στις πολιτικές παρέμβασεις και στις στρατιωτικές πολιτικές για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολυεθνικών και διαρωτώ με τέλος τι θα κάνουμε για να εμποδίσουμε το διεθνές ε, εμπόριο των διαμαντιών που έχουν εξοριχθεί και συσσωρευθεί στη διάρκεια της ε, ένοπλης σύγκρουσης. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. κύριος Φρουντζούλικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία οι αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων μας ε, καλεί να αναλάβουμε δράση αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν εκτοπιστεί, έχουν τραυματιστεί ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου και μόνο. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια διαδικασία σταθεροποίηση και οικοδομηση της ειρήνης στη χώρα αυτή. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να φέρουν πάλι τη χώρα στη σωστή τροχιά και να φροντίσουν οι πολίτες να κατευνάσουν τα πνεύματα και να αποφυπλιστούν οι παραστατικέ ομάδε. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι ροέ προσφύγων και τοπισμένων η κυβέρνηση τη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια τη ε, περιοχή, όπω τι ανισότητε ε, μεταξύ των περιφερειών τη χώρα, την ε, εξ από την εκτεταμένη φτώχεια, την ύπαρξη δικτύου διαφθοράς και την ε, ανάγκη οικονομικής ανάκαμψης. Χρειάζονται προσπάθειες από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Ευχαριστούμε κύριε μαριά για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι μια πλούσια χώρα. Έχει διαμάντια, έχει ξυλία. Και όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960. Και τα 4,5 εκατομμύρια πληθυσμός έχουν πρόβλημα. Από αυτούς τα μισή είναι παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Οι συγκρούσεις που εμφανίζονται ως θρησκευτικές συγκρούσεις στο βάθος έχουν ως υπόβαθρο την ίδια την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και κυρίως των πλούτοπαραγωγικών πηγών. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι συγκρούσεις ταυτόχρονα πολλές εταιρείες διαμαντιών και πολύτιμων λίθων έχουν άμεση σχέση με ένοπλες ομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για βιασμούς θανάτους λαιλασίες κλπ. πρέπει λοιπόν να γίνει άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να είναι πιο αποφασιστική για να σταματήσει αυτή η κατάσταση να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή και κυρίως η εκμετάλλευση των πολύτιμων λίθων και των διαμαντιών να γίνει υπέρ του ίδιου του λαού της κέντροαφρικανικής δημοκρατίας. ευχαριστώ. Κύριο Γιακόφτσης, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι μια χώρα που τα τελευταία χώρα πέρασε διάφορες διαδικασίες ε, συμφιλίωσης, ομαλοποίησης, αλλά δυστυχώς ε, η κατάσταση τον τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί σοβαρά. Μάλιστα έχουμε επιθέσεις ακόμη και στι ειρηνευτικές αποστολέ και πολλές δολοφονίες τις τελευταίες εβδομάδες. Το θέμα είναι οι βουλευτικές εκλογές θα λύσουν το πρόβλημα. Σίγουρα θα πρέπει να είναι δημοκρατικές και αν όντως γίνουν με άμεπτο τρόπο και γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα θα μπορέσουν οι βουλευτικές εκλογές με την έκβασή τους να χαράξουν τον δρόμο για την επίλυση των προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως πολλά άδειλα συμφέροντα γιατί είναι τεράστιος ο φυσικός πλούτος της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, η φυσική πόρη, ξυλία και διαμάντια κυρίως θα μπορέσει η κεντροαφρικανική Δημοκρατία να λύσει το πρόβλημα ή θα πρέπει απλώς να συνεχίσουμε τη μόνιμη μας δέσμευση με τις χώρες αυτές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και άλλες. Ευχαριστούμε κύριο Καστάλιντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι μια χώρα από το 2014 έχανα τη ζωή του ένα παιδί τη μέρα. 15.000 έχουν εκτοπιστεί από τις ε, αντιπαρατεθέμενες παραστατικές οργανώσεις. Από το 1960 η χώρα αυτή βρίσκεται σε μια κατάσταση αστάθειας και πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως λόγω των εθνοτικών και θρησκευτικών διαχωρισμών, αλλά κυρίως εξαιτίας του, νέα της νέας οικονομικής απεικιοκρατίας, που σε μια χώρα με έλλειψη δικτύου μεταφορών, οι πολίτες δεν μπορούν να φτάσουν, οι τραυματίες δεν μπορούν να φτάσουν στα νοσοκομεία, ε, που έχει σοβαρά προβλήματα. Όσο πιο πολλού πόρου έχει μια χώρα, τόσο πιο φτωχοί είναι οι πολίτε τη στην Αφρική. Ιδίω με την ξυλία που είναι τόσο πολύτιμη και την εκμετάλλευση από τι ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ. Τα διαμάντια αλίμονο δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα συμφιλίωση που έχουν προτείνει και εγκρίνει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμω ε, πολυάριθμε πράξει βία από του στρατιώτε και από ειρηνευτικέ διεθνεί δυνάμει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να τους αφοπλίσουμε. Θα πρέπει να αναλάβει ε, δράση η διεθνή κοινότητα. Γιατί δύσκολα θα έχουμε αξιόπιστες εκλογές εκεί στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίζουμε την υιοθέτηση του νέου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα νέα φαινόμενα βίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει ρητά την βιευτή όπως άλλωστε τονίζει και η δήλωση της ΥΠΑ εκπροσώπου στις 28 Σεπτεμβρίου. αυτή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις πράξεις εντός και εκτός χώρας πρέπει να λογοδοτήσουν. Και πάλι στόχος ήταν εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Ζητάμε λοιπόν να γίνει σεβαστό και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα θύματα των τελευταίων αυτών ημερών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας αξίζουν και απαιτούν ένα τέλος στις συγκρούσεις και του διαχωρισμού μεταξύ των κοινοτήτων στην χώρα. Τη στιγμή κατά την οποία η χώρα πλησιάζει στο τέλος της μεταβατικής περίοδου, τα γεγονότα θα δείχνουν πως οι εκλογές, η συμφιλίωση και η ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνουν η προτεραιότητά μας για τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να επαναλάβω την στήριξη της Ένωσης για τις μεταβατικές αρχές. Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ την Κάθριν Σάμπα Πάνσε, τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ε, μεταβατική διαδικασία. Πρέπει να συνεχιστεί η εκλογική διαδικασία, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να έχουμε ένα επίπεδο συμπερίληψης των πάντων, διαφάνειας και αξιοπιστίας που θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα αποδεκτό από όλους. Μια νόμιμη κυβέρνηση την οποία θα στηρίζει η πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό πρέπει να πάει χέρι με χέρι με τις νέες προσπάθειες για αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Η ασφάλεια είναι επίσης μια άλλη προτεραιότητα όχι μόνο ενώπιση των εκλογών. Η κεντροαφρικανική δημοκρατία εξακολουθεί να είναι ένας πολύ επικίνδυνος τόπος. Δεν πρέπει να ανεχθούμε κανέναν ο οποίος δεν τηρεί την συμφωνία αφοπλισμού και κατάπαυσης του πυρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς δικαιοσύνη. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανθρωπιστική κρίση που επηρεάζει πάνω από το μισό πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Επιπλέον, οικοδομεί γέφυρες ε, μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτός είναι ο στόχος του Ταμείου του Μπεγκού που έχει μέχρι στιγμής 108 εκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους εταίρους της ε, σκοπεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Τέλος, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία της. Μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Βεβαίως απαιτείται καλή βούληση και αποφασιστικότητα από τους ηγέτες στο Μπαγκουί και από την διεθνή κοινότητα. Άρα είναι σημαντικό να παραμείνει η κεντροαφρικανική δημοκρατία στο διεθνές προσκήνιο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Η σημερινή συζήτηση είναι μια συγκεκριμένη συνεισφορά για να μην γίνει μια ξεχασμένη κρίση κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εφτά προτάσεις ψηφίσματος έχουν υποβληθεί για το θέμα αυτό. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση.